το υλικό που θα έχουμε θα λάβουμε σύντομα τις δέουσες αποφάσεις. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα μπορούμε να κλείσουμε τη συζήτηση για το θέμα αυτό. Και συνεχίζουμε με την έκθεση του Malcolm Harbour σκάφη αναψυχής και ατομικά σκάφη. Ο πρώτος ομιλητής, ο κύριος Χάρμπορ, για τέσσερα λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που με καλέσατε να παρουσιάσω αυτή την σημαντική έκθεση για την ενιαία αγορά και θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη της Επιτροπής μας για την βοήθεια σε αυτήν την πρόταση Βλέπω εδώ τον Άντρις Φάμπερς, ο οποίος έπαιξε σημαντικό ρόλο επειδή η εκλογική περιφόρεια έχει ε, υδάτινα ε, σύνορα και πάρα πολλά σκάφη αναψυχής. Καμιά φορά πολλοί λένε γιατί χρειαζόμαστε κανονισμούς, γιατί χρειαζόμαστε εναρμονισμένους κανονισμούς για προϊόντα. Νομίζω ότι πρώτα απ' όλα είναι σημαντικό να θυμόμαστε πόσο ε, σημαντικός είναι ο μεταπητικός τομέας για τα σκάφη αναψυχής. Περιλαμβάνονται πάρα πολλοί κλάδοι και είναι περίπου 37.000 εταιρείες. Έχει γίνει πολύ καλή πληροφόρηση και έχουν επικαιροποιηθεί τα στοιχεία αυτά. Δημιουργούνται ε, πολλές θέσεις εργασίας, όχι μόνο για τους κατασκευαστές, αλλά και για τους κατασκευαστές κινητήρων θαλασσίων κινητήρων. Αυτό που προσπαθήσαμε να επιτύχουμε με εργασία νέας αγοράς είναι να προσθέσουμε αξία, να δημιουργήσουμε αυτήν την ενιαία αγορά που είναι τόσο σημαντική για τους κατασκευαστές. Αυτό που είναι ενδιαφέρον στην περίπτωση αυτή είναι ότι είναι μια πρόταση που έχει ένα μακρύ ιστορικό. Από το 1994 επικαιροποιήθηκε το 2003 και το έργο μας αυτή τη φορά ήταν να επικαιροποιήσουμε την κατάσταση για να αντιμετωπίσουμε μερικά θέματα κατά τεμαχισμού που υπάρχουν ε. διότι ε, πολλά σκάφη ε, δεν έχουν την πιστοποίηση, αλλά θα πρέπει να ασχοληθούμε με θέματα ασφαλείας και θέματα περιβάλλοντος επίσης. Απλώς για να σας ε, δείξω ε, την εμβέλεια, την σημασία του θέματος. Έχω στοιχεία από την βισκετική βιομηχανία σκαφών που ε, συμμετείχε στις διαβουλεύσεις που οδήγησαν σε αυτήν την πρόταση και από ό,τι μου είπανε αυτές οι νέες υποχρεώσεις αυξάνουν την ασφάλεια και έχουν ωφέλη περιβαλλοντικά και θέτουν τέρμα ε, στις εθνικές διαφοροποίησεις που κατατεμαχίζουν την αγορά ε, και αναγκάζουν τους κατασκευαστές να προσαρμόσουν την κατασκευή. Είναι σημαντικό να έχουμε μια ενιαία αγορά και καμιά φορά ξεχνούμε ότι ε, σε με μικρά βήματα δημιουργούμε ένα σημαντικό οικονομικό χώρο, ε, μια ολόκληρη αλυσίδα εφοδιασμού ευρωπαϊκή που είναι κάτι καλό για τους ε, καταναλωτές, ε, για το περιβάλλον και για τους παραγωγούς. Ποια είναι τα βασικά σημεία. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ότι η αποδοτικότητα η περιβαλλοντική των κινητήρων είναι κάτι σημαντική, όπως ε, με άλλους κινητήρες εσωτερικής καύσης αυτοί θα βελτιωθούν. Η Κομισιό ήταν αρκετά οξυδερκής διότι ευθυγράμμισε τους κανονισμούς με τις Ηνωμένε Πολιτείες, τόσο ώστε να έχουμε έναν κλάδο παγκόσμιο. Επίσης επιφέραμε λεπτομερείς αλλαγές ταξινόμηση ε, των ε, σκαφών, των ατομικών σκαφών αυτό δεν ήρθε από την Κομισιόν, αλλά θα ήθελα να ευχαριστώ την Κομισιόν γιατί δέχθηκε τις αλλαγές. Κάναμε τη δική μας αξιολόγηση αντικτύπου για την πρόταση που μπορούμε να παρουσιάσουμε στο Συμβούλιο και, ε, και λειτουργήσε αυτό και στην περίπτωση που κανείς σκεφτεί ότι είναι αυτό με ένα μέσο ε, σκοτεινό. Θα δείτε τι επιρροή έχουν αυτές οι αξιολογήσεις. Υπάρχουν άλλες λεπτομερείς αλλαγές και είμαι ε, βέβαιος ότι θα ασχοληθούμε αργότερα όταν απαντήσω στο τέλος της συζήτηση. Με μεγάλη ευχαρίστηση σας παρουσιάζω αυτή την πρόταση. Υιοθετήθηκε ομόφωνα από την Επιτροπή μου και ελπίζω ότι θα τύχει της ίδιας αντιμετώπισης αύριο εδώ στην ψηφοφορία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Χάρμπορ. Και τώρα θα ήθελα να δώσω τον λόγο στον Επίτροπο Ταγιάννη. Κύριε Πρόεδρε, Αξιότιμοι κύριοι Ευρωβουλευτέ, καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω το σώμα και όλος ιδιαιτέρω τον πρόεδρο Χάρπορ που είναι εισηγητή τη πρόταση που επέτρεψε την εξέβρεση συμφωνία για αυτό το κείμενο οδηγίες για τα σκάφη. Ε, κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης μιλήσαμε ιδιαίτερα όσον αφορά τον περιορισμό των εκπομπών ε, από τα σκάφη αυτά και εισήγαμε και πιο, αυστηρούς, ε, πιο αυστηρά όρια, αλλά θελήσαμε να θέσουμε τα σκάφη αυτά στο τελευταία νομοθετική ρύθμιση και αυτό αφορά τις υποχρεώσεις, τους κοινοποιημένου οργανισμούς και τους εμπλεκόμενους φορείς. Οι βασικές αλλαγές βελτιώνουν την προστασία του περιβάλλοντος και τον τομέα των, λιμένων, των ε, λιμένων σκαφών αναψυχής. Ε, μειώνονται κατά 25% οι αιτήσει εκπομπές ε, οξυδίου του αζότου και ε, υδρογοναθράκων από τα σκάφη αυτά. Για να εγγυηθούμε τη σύνδεση ανάμεσα στις διάφορες πρωτοβουλίες, υιοθετήσαμε μια στρατηγική που πέρα από την προστασία του περιβάλλοντος έχει την ε, ιδιαιτερότητα ότι προωθεί την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής ε, ε, βιομηχανίας και θέλω να υπογραμμίσω πόσο σημαντικό είναι αυτό ο τομέας γιατί υπάρχουν 37.000 επιχειρήσει με πάνω από 230.000 εργαζόμενους 90 ε, δις ε, τζίρο έκανε το 2011 και οι περισσότερες είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, στην Ευρώπη έχουμε 48 εκατομμύρια ανθρώπους που κάνουν αναψυχή και με σκάφη και χρησιμοποιούν σκάφη με κινητήρες ή με ιστία. Μιλάμε για τεράστια μεγέθη δηλαδή. Επίσης ευθυγραμμίσαμε τα όρια εκπομπών με αυτά των ΙΠΑ. Προτείναμε και ένα μηχανισμό μεταβατικό για να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να προσαρμοστούν στους κανόνες εκπομπών που είναι πιο αυστηροί. Το η δέσμη μέτρων για την οποία συζητάμε σήμερα είναι κατά τη γνώμη μου ένα εξαίρετο παράδειγμα ε, παντρέματος ανάμεσα στη βιομηχανική και την περιβαλλοντική πολιτική που πρέπει να προωθούμε όλο ένα και περισσότερο στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στηρίζοντας την ανταγωνιστικότητα του βιομηχανικού μηχανικού συστήματος όσον αφορά τώρα τις κατηγορίες ε, των διαφόρων των ε, λουωμένων έχουμε διάφορες ε, κατηγορίες και αυτό γιατί οι κατασκευαστές αλλά και οι χρήστες έχουν διαφορετικές συνήθειες Έχουμε να δούμε τον αντίκτυπο στους κατασκευαστές και τις συνέπειες στους, κατα... Ε, καταναλωτές. Δεν είμαστε αντίθετοι για αναθεώρηση των κατηγοριών ε, για, τις... Ε, για τα διάφορα είδη σκαφών, αλλά θα πρέπει να γίνουν εις βάθος μελέτες και αυτό δεν μπορεί να γίνει σε μια νυχτή. Γι' αυτό αποφασίσαμε να αφήσουμε το σημείο αυτό ώστε να αντιμετωπιστεί στην επόμενη εξέταση της οδηγίας για τα σκάφη, σκάφη αναψυχής. Επίσης, δεχτήκαμε και την πρόταση του Κοινοβουλίου που τροποποιεί την διατύπωση των ε, υφιστάμενων ε, ε, κατηγοριών. Όσον αφορά το όριο εκπομπών, ακουστικών εκπομπών, θεωρήσαμε πως δεν χρειάζεται να το αλλάξουμε αυτή τη στιγμή, γιατί οι ενοχλήσεις που προέρχονται από τα σκάφη ψυχής οφείλονται σε διάφορα πράγματα. Ωστόσο, το ότι μπορούμε να μετρήσουμε την επιρροή χωρίς να αλλάξουμε τα σκάφη σύμφωνα με την οδηγία. Ε, ε, ε, διευκρινίσαμε αυτή την αναλλακτική στο άρθρο 5 και έπειτα αποφασίσαμε να συμπεριλάβουμε για την, στις για την επόμενη ενημέρωση της οδηγίας και τα όρια εκπομπών αερίων αλλά και θορύβων. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε τα αποτελέσματα των εργασιών που θα ξεκινήσουμε στο μέλλον, αλλά σίγουρα θα εξετάσουμε προσεκτικά τη δυνατότητα ε, νέων προόδων στο πλαίσιο της προστασίας του περιβάλλοντος και θα λάβουμε υπόψη όλες τις απαιτήσει ανάπτυξης και απασχόλησης με ιδιαίτερη προσοχή στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. ευχαριστώ πολύ, Επίτροπε. Και τώρα θα ήθελα να δώσω μέσα στο λόγο στον κύριο Ταταρέλα. καλό δεν τον βλέπω στην αίθουσα. Επόμενο ο μιλητής τότε, ο κύριος Σφάμπ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε ε, Πρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής, θα ήθελα καταρχάς να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο της Επιτροπής μας, κύριο Χάρμπορ. Έχει κάνει εξαιρετική δουλειά για τα σκάφη ε, αναψυχής και να μην ξεχνάμε και τα, ε, τις μηχανές, τα jet ski που κυκλοφορούν ε, στο νερό. Επίσης, ε, τα ανέφερε και ο ίδιος, ε, αυτό που μας ενδιαφέρει κυρίως είναι η καλή πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι ε, και ευρωπαϊκή πρόταση για την ευρωπαϊκή αγορά να να την υποστηρίξουμε. Γιατί ε, ευτυχώ μπορεί κανεί παντού στην Ευρώπη και στη θάλασσα και στι λίμνες και στα ποτάμια να χρησιμοποιεί και γερμανικά και ιταλικά σκάφη και καλό είναι έτσι λίγο να το ομοιονοποιήσουμε έτσι ώστε και οι κατασκευαστέ και οι ε, χρήστε να έχουν μια ευρωπαϊκή υπεραξία. Ένα δεύτερο που καταφέραμε να ξεκαθαρίσουμε και ευχαριστώ πολύ είναι οι εκτιμήσει επιπτώσεων και ε, που ζητάει το Κοινοβούλιο να έχουν και μια πρακτική χρηστικότητα. Δηλαδή, όταν είναι καλοί οι και επιστήμονε που μπορούν να κάνουν αυτέ τι ε, μελέτε επιπτώσεων και τελικά να πιστούν οι συνομοθέτε ότι ο δρόμο που προτείνουμε ε, είναι ο δρόμο προ τη λύση. Και αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Αντιπρόεδρε τη Επιτροπή, κύριε Πρόεδρε, η πρόταση για τη μελέτη σκοπιμότητας δείχνει με καταπληκτικό τρόπο ότι με αυτή τη τεχνική δουλειά βοηθούμε τους πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους προσθέτουμε μια ευρωπαϊκή αξία. Ως νομικός επίσης το βλέπω και από τη νομική σκοπιά. Τώρα βρέθηκε μια συνένεση στην Επιτροπή, ομόφωνα μάλιστα, και έχουμε την ασφάλεια ότι τα σκάφη αναψυχής αλλά και τα jet ε, θα εγγραφούν στη συνθήκη της Σαββόνας και θα ανταποκρίνονται στη νέα νομική πραγματικότητα ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει την ίδια δήλωση στην οδηγία για τα πυροτεχνήματα. Ε, Παρ' όλα αυτά, ελπίζω αύριο να υποστηριχθεί η πρόταση αυτή με μεγάλη πλειοψηφία. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Ρέπο, για ένα λεπτό. Ναι. Υπήρξε, ήταν με μεγάλη χαρά και τιμή που ήμουν σκιώδης εισηγητής για την ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών για το θέμα των σκαφών αναψυχή και ατομικών σκαφών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Χάρμπορ για καλή συνεργασία. Κάτω από τη δική του διεύθυνση μπορέσαμε να έχουμε μια εξαίρετη έκθεση για να προωθήσουμε την προστασία των καταναλωτών και την αηφόρο ανάπτυξη. Από την άποψη των καταναλωτών βελτιώνεται σημαντικά η ασφάλεια εχνήλαση των οχημάτων, πρόληψη ατυχημάτων, όταν ε, τα οχήματα ή τα σκάφη αναποδογυρίζουν και έχουμε επίσης ε, των ηλεκτρονικών ε, συστημάτων ε, και των κινητήρων με αέριο που προστατεύονται. Επίσης τα βιοκαύσιμα προωθούνται και χαίρομαι που αυτή η μεταρρύθμιση υποστηρίζει τους επιχειρηματίες των τομέα των σκαφών και μας οδηγεί σε μια ασφαλέστερη και πιο αηφόρο Ευρώπη. Ο κύριος Μάντερ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα είμαι σύντομο. Θέλω να ευχαριστήσω ειλικρινά τον Μάλκομ Χάρμον για την εντατική συνεργασία της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και δείχνει η ομόφωνη έγκριση της έκθεση ε, πόσο σπουδαία δουλειά έχει κάνει. Συχνά αμφιβάλλω εγώ για τις εκθέσεις ε, ε, που στέλνουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ταξινομούνται κάθετα προς τον κάθελαθο των αχρήστων δηλαδή και δεν αξιοποιούνται. Αλλά χαίρομαι τώρα που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε ε, την έκθεσή μας και πιάνει τόπο. Η ασφάλεια για τους χρήστες και για το περιβάλλον βελτιώνεται και είναι και ε, πραγματικά πολύ ε, καλή αυτή η προσπάθεια για τους χρήστες και των ε, σκαφών αψυχής και των δικύκλων στη θάλασσα ε, θα πρέπει να έχουμε ε, και ένα ευρωπαϊκό πλέον δίπλωμα έτσι, για να οδηγεί κανείς αυτά τα σκάφη. Δεν αρκεί να είναι τα σκάφη από μόνα τους ασφαλή, θα πρέπει και οι οδηγοί τους να έχουν την κατάρτιση. Δεν ξέρω τι φρονεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά. Αύριο πραγματικά θα ψηφιστεί και θα εγκριθεί με μεγάλη πλειοψηφία αυτή η έκθεση και βοηθούμε και βελτιώνουμε κατά την ε, αγορά. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα για ένα λεπτό η κυρία Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επίτροπε Ταγιάννη, συνάδελφοι. Πολλά Συγχαρητήρια στον φίλο Πρόεδρο Χάρμπορ για την εξαίρετη του εργασία για την ασφάλεια των σκαφών αναψυχής και την προστασία του ε, περιβάλλοντος. Είναι πολύ σημαντικό θέμα προφανώς για την Ιταλία, αλλά το ίδιο σημαντική είναι και η προστασία της ασφάλειας των όσων σε αυτή την ίδια θάλασσα δεν χρησιμοποιεί σκάφος, αλλά κολυμπά. Στη χώρα μου κάθε χρόνο σκοτώνονται ένα σωρό άνθρωποι από τις έλικες των ίδιων αυτών σκαφών αναψυχής χωρίς καν αυτοί να το, οι οδηγοί των σκαφών να το αντιληφθούν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να καταστεί υποχρεωτικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στρέφομαι στον ε, στον Επίτροπο, ώστε να υπάρχει απαγόρευση ε, να φτάνουν τα σκάφη αυτά πέρα από το, πιο κοντά από τα 50 μέτρα ε, από την παραλία, για ώστε να προστατεύονται οι λουόμενοι. Ευχαριστώ. Κυρία Χάνσλεκ, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, αξιότιμοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Θέλω να συγχαρώ εκ βάθους καρδίας τον εισηγητή μας. Έχει κάνει καταπληκτική δουλειά και πολύ καλούς συμβιβασμούς. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε μερικά εκατομμύρια σκάφη αναψυχής. Και κανονικά ε, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλες οι προδιαγραφές και οι απαιτήσει ασφαλείας που ισχύουν σήμερα η πρόταση ευρωπαϊκή Επιτροπής προσαρμόζει την κείμενη νομοθεσία σε προδιαγραφές ασφαλείας και σε περιβαλλοντικά κριτήρια. Μεταξύ αυτών είναι και η χορύπανση αλλά και η εκπομπή καυσαερίων. Είναι πολλά τα είδη των σκαφών, δεν είναι μόνο σκάφη πλοία δηλαδή, αλλά ε, και γιότ και ιστιοφόρα και εξολέμβια, αλλά και πολύ ε, μικρότερες ακριβώς ε, βάρκες εξολέμβειες Ο καουτσούκ ε, και θα πρέπει πραγματικά να ανταποκρίνονται σε όλα τα κριτήρια ασφαλείας ε, και θα πρέπει να τονίσουμε ότι στο τομέα των σκαφών αναψυχής είναι πάνω από 37.000 οι εταιρείε που δραστηριοποιούνται, εκ των οποίων πολλές μικρομεσαίες. Ε, και ε, ε, είναι πάνω από 270.000 οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις αυτές. Οι εταιρείε αυτές και οι εργαζόμενοι θίγονται, λοιπόν, μάλλον τους αφορά αυτή η νέα ρύθμιση. Συγχαρητήρια και πάλι στον εισηγητή. Στην Επιτροπή ΙΜΚΟ κατάφεραν ε, πολλά να βελτιωθούν, να ξεκαθαριστούν ιδιαίτεροι ορισμοί. Είναι πολύ τεχνική δουλειά και ευχαριστώ πολύ τον Μάλκομ Χάρμπορ και τον συγχαίρω. Μπράβο σου και πάλι, ειλικρινά, σου εύχομαι καλή επιτυχία στη συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Next speaker is Mr. Ο Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας, τον Μάλκομ Χάρμπορ, για την πρόταση αυτή και την τόσο σημαντική έκθεση. Έχουμε ξαναδεί ανάλογα ψηφίσματα στο Κοινοβούλιο, ε, αλλά η συγκεκριμένη έκθεση είναι πραγματικά πάρα πολύ καλή για να συστηματικοποιηθεί λίγο ε, ο κλάδος. Και θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή στο εξής χρειαζόμαστε προδιαγραφές ε, που όμως να μην ε, επιτρέπουν μονοπόλια των μεγάλων κατασκευαστών. Θα πρέπει και οι μικροί και οι μεσαίοι να έχουν πρόσβαση σε αυτή την αγορά ε, για μικρά σκάφη αναψυχής και Είμαι πεπισμένος ότι η πρόταση αυτή θα αποτελέσει ένα σαφές μήνυμα για καλύτερη ρύθμιση του κλάδου. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Κάλπελτς, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Να ευχαριστήσω και τον πρόεδρο της Επιτροπής ΣΥΜΚΟ και να το συγχαρώ για την έκθεσή του. Είναι πραγματικά κάτι που του αξίζει, διότι η έκθεσή του ψηφίστηκε ομόφωνα στην Επιτροπή, προσθέτει ευρωπαϊκή αξία, έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, πάρα πολύ επιμελή και εμπεριστατωμένη, έχει βγει σε πολλές λεπτομέρειες και τεχνικές και τις διευκρινίζει και έχει λύσει και προβλήματα. Θέλω να τονίσω τα εξή εγώ. Δεν έχω και πολύ χρόνο. Οι οριακές τιμές πρέπει να εναρμονιστούν. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο αυτό και απαραίτητο. Αν δούμε τις τεχνολογικές εξελίξεις και ε, τις νέες προδιαγραφές και προσπαθήσουμε να τις υποστηρίξουμε, θα είναι προς όφελος όλων, ιδιαίτερα ε, εάν αυτές οι προδιαγραφές γίνουν και παγκόσμιες ταυτόχρονα. Ε, ένα δεύτερο στοιχείο, οι ροικές τιμές και για τις εκπομπές ρήπων ε, ή για την ηχορή, πανσήμιωση του θορύβου, δηλαδή σιγαστήρες και ε, περιορισμός της ταχύτητας είναι κάτι επίσης πολύ χρήσιμο. Ένα δεύτερο θέμα που θέλω να αναφέρω έχει να κάνει με τη ρήτρα ασφαλείας. Θα ήθελα να πω ότι επιτέλους έχουμε μια νομική βάση για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και στην απόσυρση κάποιων σκαφών ή κάποιων κινητήρων που συνιστούν απειλή για τους λουωμένους ή γενικότερα για τη δημόσια υγεία. Επίσης, θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να αρχίσουν οι νέες διαδικασίες αξιολόγησης πλέον να ισχύουν, ιδιαίτερα τη στιγμή που οι περισσότεροι ε, χρήστες αγοράζουν ε, τα σκάφη αυτά από τρίτες χώρες που δεν ανταποκρίνονται στις δικές μας προδιαγραφές. Τουλάχιστον μέχρι τώρα αυτό δεν ίσχυε. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί ε, στη δράση μας, μεθοδικοί, γιατί είναι πολλοί οι χρήστες. Ο πρόεδρος διακόπτη. Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής, ο κ. Κονφεράτη, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, το θέμα που συζητάμε αποτελεί μια εξαιρετική πρόταση οδηγίας ε, για τα ε, σκάφη αυτά. Ευχαριστούμε τον κύριο Σιγητή αλλά και τους Σκιώδης και ευχαριστούμε και την Κομισιόν που έδωσε ιδιαίτερη προσοχή σε ορισμένες σημαντικές πτυχές. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να συμπληρωθεί αυτή η οδηγία με τον προσδιορισμό των κατηγοριών ε, σχεδιασμού. Με τόσα είπατε κι εσείς εδώ, αλλά αυτό που μου φαίνεται σημαντικό μπορεί να είναι ένα σημείο αναφοράς και ένα μικρό μοντέλο και είναι το ότι έχει επιλεχθεί για αυτό το τομέα το θέμα της ασφάλειας και του σεβασμού του περιβάλλοντος, όχι μόνο ως αξίες για τους χρήστες και επομένω για τους καταναλωτές, αλλά και ως κεντρικό άξονα για ένα μοντέλο ανταγωνιστικότητας που σε αυτό το τομέα αφορά τις μικρές και μέσες επιχειρήσεις και θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε πάρα πολλού ε, κλάδους. Ε, είμαι σίγουρος ότι αύριο θα εγκριθεί η πρόταση, αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε αυτές τις δύο πτυχέ στο περιβάλλον και η ασφάλεια μαζί καθιστούν δυνατό έναν ανταγωνισμό υψηλού προφίλ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και τώρα θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία Κατσιάη. Έχω μόνο έναν ομιλητή, τον κύριο Πάσκα, για ένα λεπτό. Ε, Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, τα διάφορα ε, σκάφη ε, μπορεί να δημιουργήσουν θέματα περιβάλλοντος ε, και άλλα προβλήματα. Πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε Πρέπει να εκτιμήσουμε ιδιαίτερα το έργο όλων όσων συμμετείχαν στην έκθεση αυτή. Η οδηγία καλύπτει όλα τα σκάφη ε, από τα μικρά μέχρι τις μεγάλες θαλαμιγούς και θα έπρεπε να βρεθούν κοινέ απαιτήσει που πρέπει να φροντίζουμε να τηρούνται. Η ασφάλεια του κινητήρα, των, ηλεκτρικών, των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, ε, και η επίδραση των εκπομπών, ρήπων αυτών των σκαφών ε, πρέπει να εξετάζονται. Είμαι πεπισμένος ότι οι νέες αυτές ε, διαδικασίες ε, θα βελτιώσουν την διαδικασία αξιολόγηση όλων των ε, σκαφών. Και τώρα ο Επίτροπος Ταγιάννη. Έχετε τον λόγο, Επίτροπε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους τους βουλευτές ε, που συνεισφέραν στο να πετύχουμε ένα τόσο σημαντικό αποτέλεσμα για την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και για μια σύγχρονη και ανταγωνιστική βιομηχανική πολιτική. Συμφωνώ με τον κύριο Κοφεράτη εδώ. Το μήνυμα αυτό το δίνουμε και για το μοντέλο της ανάπτυξης και για μια βιομηχανική πολιτική που να μην μολύνει αλλά και να είναι και πρωταγωνιστική στον τομέα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Άκουσα επίσης ενδιαφέρουσες προτάσεις ε, του κ. και του κ. Ντεμαρτίνη. Θεωρώ ότι είναι πολύ καλές ε, ιδέες να εξετάσουμε ε, ακριβώς το θέμα του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Έχω ζητήσει ήδη στη Γενική μου Διεύθυνση να αξιολογήσει την δυνατότητα και την καταλληλότητα να προετοιμάσουμε μια τέτοια πρόταση, όμως ε, δεν έχουμε βρει τη νομική βάση στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς για το οποίο είμαι υπεύθυνο αλλά θα μπορούσε να βρεθεί μία νομική βάση στον τομέα των μεταφορών όπου ήδη υπάρχει ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ε, για τα ε, σκάφη μεταφοράς εμπορευμάτων ή επιβατών στις ερωτερικές πλωτές οδούς. Έτσι λοιπόν θα ζητήσω από τη Γενική Διεύθυνσή μου να έρθει σε επαφή με τη Γενική Διεύθυνση του Αντιπρόεδρου Κάλλας για να εξετάσουμε ακριβώς τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε ένα τέτοιο ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας το ίδιο ισχύει και σε ό,τι αφορά ε, αν, ό,τι αφορά την εξέβρεση μιας λύσης ευρωπαϊκής ε, για το BOE. Και εγώ νομίζω ότι πρέπει να δούμε τις ε, πληροφορίες που έχουμε συλλέξεις. Ό,τι αφορά το συμβιβαστικό πακέτο, εμείς είμαστε θετικοί απέναντι στο σύνολο, θέλουμε γρήγορη υιοθέτηση. Παρ' όλα αυτά έχουμε κάποιες αμφιβολίες σε σχέση με την αρμοδιότητα ε, της Επιτροπής ε, που ιδρύει η οδηγία και έχουμε διαβιβάσει στο Κοινοβούλιο μια σχετική δήλωση για τα πρακτικά της Ολομέλειας. Ευχαριστώ επίσης τον κύριο Χάρμπορ εκ και όλα τα μέλη του Κοινοβουλίου που μας ε, επέτρεψαν να δώσουμε ένα θετικό μήνυμα σε ένα τομέα που αντιμετωπίζει κάποιες δυσκολίες, όμως τέτοια μηνύματα ε, έχουν ως αποτέλεσμα να ενθαρρύνουν τη βιομηχανία και τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι οι μόνες σήμερα που μπορούν να δημιουργήσουν αίσθηση εργασία και να δώσουν κάποια ελπίδα και στους νέους μας. Σα ευχαριστώ. Thank you very much, Ευχαριστώ, Επίτροπε. Και εν τέλει θα ήθελα να ζητήσω από τον εισηγητή, τον κύριο Χάρμπορ, να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω όλους τους προλαλήσαντες συναδέλφους που συνέβαλαν και ήταν πάρα πολύ ευγενείς προς το έργο μου. Ε, είναι μια, ένα, κοινό έργο πρέπει να ομολογήσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Βλέπω ότι όλοι οι σκιώδεις ε, έχουν εξαφανιστεί, διότι βέβαια έχουμε προχωρήσει ε, σήμερα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Σφάμπ, ανέφερα τον κύριο Ρέπο, τον κύριο Μάντελς και την ε, ε, κυρία Ρούλερ από τους Πράσινους που δούλεψε πολύ σκληρά. Καλύψαμε μερικές από τις πτυχές. Θα ήθελα να σκεφτούμε ότι τώρα είμαστε στο στάδιο υλοποίησης. Είχαμε συζητήσεις επίπονες και πολλά από τα θέματα που συζητήσαμε στην Επιτροπολογία. Θα ήθελα να ακούσω την ε, τελευταία άποψη της Επιτροπής για την συμβαστική πρόταση, αλλά θέλουμε το Κοινοβούλιο να συνεχίσει να παρακολουθεί αυτό που συμβαίνει. Δεν έχουμε ένα συγκεκριμένο ρόλο στις διαδικασίες υλοποίησης, αλλά πιστεύω ότι δεν είναι ικανοποιητικό απλά να περνάμε νομοθεσίες και μετά να μην βλέπουμε πώς υλοποιούνται στην πράξη, ιδιαίτερα λόγω του χρόνου που μεσολαβεί από αυτές τις τροπολογίες. Εγώ ε, για την Επιτροπή μου και για τη ε, διαδοχή ε, πιστεύω ότι θα πρέπει να παρακολουθηθεί και έχουμε για μελλοντικές ενισχύσεις όπως την περιβαλλοντική απόδοση, τις εκπομπές ρήπων και θορύβου. Περνά χρόνος από την ψηφοφορία που ήταν πέρσι τον Ιούνιο μέχρι να φτάσει αυτό στο Κοινοβούλιο. Και αυτό γιατί οι δικοί στο Συμβούλιο οι... δεν συναντιούνται τόσο συχνά. Ε, και αντί να επιστρέψουμε μια δεύτερη ανάγνωση θα του στέλναμε την πρώτη μα ανάγνωση και όλα τα στοιχεία και τις ε, αξιολογήσει αντικτύπου και μετά να συγκροτήσουμε ένα τελικό πακέτο. Αυτό έγινε κατά τη διάρκεια της Ιλλανδικής ε, προεδρία και ήθελα να ευχαριστήσω τον Μάικλ Κλάιν που ήταν επικεφαλή μαζί με τι υπηρεσίε τη Κομισιόν και του συναδέλφου που κατέληξαν σε αυτή τη συμφωνία. Αυτό κλείνει αυτή τη διαδικασία. Προσβλέπω προ μια θετική ψήφο αυτή την πρώτη πρόταση αύριο. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρίε και κύριοι, έχει κλείσει η συζήτηση στο θέμα αυτό. Αύριο η ψηφοφορία στις 11.30. Περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο. Πρόταση ψηφίσματος, τεχνικές απαιτήσεις και διοικητικές διαδικασίες όσον αφορά